τα προνόμια και τις ασυλίες που συνοδεύουν το, την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή. Έχω λάβει από τον κύριο Βίκτορ Σπάτσιτς ε, μία αίτηση για την πράσπιση της ε, ε, βουλευτικής του ασυλίας με βάση το άρθρο 6.2 ε, θα παραπευθεί στην αρμόδια νομική επιτροπή που είναι η νομική επιτροπή. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες μου έδωσαν τον κατάλογο για τους διορισμούς στις διάφορες επιτροπές. Θα δημοσιευτούν στα πρακτικά και αν δεν διατυπωθούν ενστάσεις μέχρι την έγκριση των πρακτικό θα θεωρούν ως συγκεκριμένοι διορισμοί στην Επιτροπή ΑΦΕΤ, ο κύριος Σοφοκλής Σοφοκλέος και στην Υποεπιτροπή Άμυνας ο κύριος Σοφοκλής Σοφοκλέος. Και περνάμε στις ψηφοφορίες. Πρώτη έκθεση είναι η έκθεση του κυρίου Μπέντσεν.